przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym dziennego jest... Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Το πρώτο θέμα είναι της ημερήσιας διάταξης. Είναι η έκθεση της κυρίας Καρνιέται διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά καθώς επίσης η έκθεση του κυρίου Ντεκάμπος εν αγορά των Ευρωπαίων πολιτών εν αγορά για τις επιχειρήσεις πρόκειται για κοινή συζήτηση βεβαίως Σίλβιο Μπουσόη και δημόσια σύμβαση δήλωση της Επιτροπής εγώ απευθύνω το καλώς ορίσατε στον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ καθώς επίσης και την εκπρόσωπο της Προεδρίας, την ε, Υπουργό κυρία Γέρη. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους τρεις εισηγητές και πρώτα η κυρία Σάντρα Καρνιέτη. Madame Kalniete. Oh, ah, Mr. President, sorry. I... Με συγχωρείτε Πρόεδρε. Μέχρι να ακούσω τη μετάφραση της ε, εκφώνησής σας, καθυστέρησα. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι αν θέλουμε να πιστεύουμε στο